Έτσι λήγουν οι σημερινές μας εργασίες. Ε, μία πληροφόρηση και μόνο από το ΕΛΚ ζητήθηκε στην, στον έλεγχο προϋπολογισμού η κυρία Πέτρη Σαρβάμα, το ίδιο στην Επιτροπή Μεταφορών και στη συνεργασία Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Φαίνεται πως όχι εγκρίνονται